στην αγορή εργασίας. Το άρθρο 24 του, της χάρτας του ΟΙΕ το προβλέπει ούτως ώστε να μην αποκλείονται αυτά τα άτομα από το εκπαιδευτικό σύστημα. Τώρα, έκθεση της κυρίας Γέγλ. Ο ρόλος των γυναικών στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές. Για τέσσερα λεπτά η κυρία Γέγελ. Όχι, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ως εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για την έκθεση ε, πρωτοβουλίας ε, ο ρόλο των γυναικών στον τομέα τη γεωργίας και τις αγροτικές περιοχές ήθελα να γίνει ε, μια συζήτηση για τον πολυλειτουργικό ρόλο των ε, ε, γυναικών στις αγροτικές περιοχές. Κεντρική καθήκον της ευρωπαϊκής πολιτικής για τι αγροτικές περιοχές είναι να υπάρχουν ίσε συνθήκες για όλες τις περιφέρειες και να υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη και των αγροτικών και των αστικών περιοχών έτσι ώστε να υπάρχουν προοπτικές ο κόσμος να μείνει στην Ήπεθρο. Τις περασμένες ε, δεκαετίες η γεωργική πολιτική ε, είχε στόχο τη θετική ανάπτυξη της Ήπεθρου. Ε, θα πρέπει, θέλαμε να φτιάξουμε ένα ε, χώρο ο οποίος ε, να είναι βιώσιμος. Όμως αυτό επιζητά περαιτέρω προσπάθειες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λοιπόν το δυναμικό των γυναικών στις αγροτικές περιοχές. Η ποιότητα ζωής και η οικονομική δύναμη στις αγροτικές περιοχές μπορεί να ε, ενισχυθεί με την παρουσία των γυναικών και τη δράση τους. Έχει τα τελευταία χρόνια καταδειχθεί ξεκάθαρα ότι η υπεράσπιση των γυναικών και των σχεδίων τους ε, επιφέρει σημαντικές προόδους γενικά στην Ήπεθρο. Η εμπειρία αυτή ε, μέσα στα πλαίσια της ενίσχυσης από το δεύτερο πυλώνα ε, έχει να κάνει και με την γενικότερη ενίσχυση των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γυναίκες είναι σημαντικές στα περασμένα χρόνια οι γυναίκες ε, έχουν συμβάλει σημαντικά στην ε, ε, ποικιλομορφία της αγοράς. Οι αγροτικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα, δίνουν καινοτόμες υπηρεσίες μαζί με την παραγωγή τροφίμων. Αυτό το δυναμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο αυτή τη στιγμή ε, πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά την ε, συμβολή των γυναικών στις αγροτικές περιοχές, να λάβουμε υπόψη μας τις ικανότητές τους και τις δυνατότητές τους και τη συμβολή τους. Θα πρέπει οι γυναίκες να συμμετέχουν πλήρως στους πόρους της αγροτικής ζωής και της οικονομικής ζωής. Οι αγρότησες ε, ανάλογα με την επιχειρηματική τους ευθύνη θα πρέπει να έχουν και τα ανάλογα δικαιώματα. Θα πρέπει να ε, εκπροσωπούνται στις, ε, στα αγροτικά συμβούλια, να υπάρχει κοινωνική ασφάλεια για τις γυναίκες αυτές που εργάζονται στην Ήπεθρο. Μετά από εντατικό ε, διάλογο καταφέραμε στην Επιτροπή Γεωργίας ε, να ψηφίσουμε, να υπερψηφίσουμε την έκθεση με μόνο μία ψήφο κατά. Ε, αύριο στην ε, Ολομέλεια δεν θα κατατεθεί καμία τροπολογία. Αυτό μου δείχνει ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό συμβιβασμό που καταφέραμε να επιτύχουμε μέσα από τη συμβολή όλων των ομάδων. Αυτό σημαίνει ότι με ομοφωνία όλοι μαζί θέλουμε να δώσουμε βάρος ε, στην έκκλησή μας ε, να δοθεί και από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο αντίστοιχο βάρος σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, ειδικότερα τις κοιόδες ε, για την εξαίρετη συνεργασία μας. Η συνεχής συζήτηση για το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013 πρέπει να λάβει υπόψη το ρόλο των γυναικών στον γεωργικό τομέα. Είμαι αισιόδοξη ότι η έκθεσή μας θα αποτελέσει θεμέλιο για αυτή τη ουσιαστική και απαραίτητη συζήτηση και ότι η συνεισφορά μας θα ε, ληφθεί υπόψη και στη συνεχή συζήτηση για τα οικονομικά μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, με κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συγχαίρω την Ελίζαμπεθ Γέγκελ για την καλή εργασία στην εισήγηση αυτή και την συνεχιζόμενη εργασία και προσπάθειες κατά τη διάρκεια των ετών που τη γνωρίζω. Βεβαίως είναι σημαντικό που δεν υπάρχουν τροπολογίες που κατατέθηκαν ε, θα ήθελα να επισύρω την ε, προσοχή πάνω στην παράγραφο 4 για την ε, προϋπολογισμό για την γεωργία, παράγραφο 10 νέες τεχνολογίες στην Ήπεθρο και να διεύρυνση της πρόσβασης στα βριζονικά οι γυναίκες θα πρέπει να εκπροσωπούνται ε, σε όλα τα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά σώματα ε, στον αγροτικό τομέα, ούτω ώστε να βλέπουμε και τις ε, δύο πλευρές, τους άνδρες και τις γυναίκες. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρες στον τομέα αυτό και θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό και θα πρέπει η Κομισιό να συνειδητοποιήσει ότι τα πρόβλημα για τους αγρότες και τις αγρότησες θα είναι στο επίκεντρο της συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική της μεταρρυθμίσης και θα χρειαστούν ίσως περισσότερες δαπάνες. Θα ήθελα να διαβιβαστεί το μήνυμα αυτό στην Επιτροπή. Η κυρία Τικάου. κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η βασική επιδίωξη των γυναικών είναι να βρουν εργασία στον αγροτικό τομέα και έχουμε μειωμένες αποδοχές για τους ηλικιωμένους. Επίσης η εκπαίδευση, η σταθμή, η βρεφονιπιακή είναι σημαντική. Η επισφάλεια στον αγροτικό τομέα μειώνει την ενδιαφέρον ε, των επιχειρηματιών για εκμεταλλεύσεις παραγωγικές στον τομέα αυτό. Θα πρέπει τα διαρθρωτικά ταμεία να καλύψουν ε, το κενό, την έλλειψη των υποδομών και να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων στις υποδομές αυτές. Θα πρέπει να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας να διευκολύνουμε την πρόοδο του διαδικτύου στις αγροτικές περιοχές, να δημιουργηθούν επίσης θέσεις εργασίας συνδυάζοντας ε, την οικογενειακή ζωή με τις επαγγελματικές δραστηριότητες ενθαρρύνοντας έτσι ε, τους αγροτικούς πληθυσμούς να παραμείνουν ε, στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Γέγκλο και να την ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία. Βεβαίως, έχουμε ε, στις 3 ε, στις δέκα εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις ε, διευθύνουν οι γυναίκες. Θα πρέπει να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές ούτως ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην γεωργία, να διευκολυνθεί η καθημερινή του ζωή με υπηρεσίες όπως φροντίδα, εκπαίδευση, διάφορες ψυχαγωγικές ασχολίες. Θα πρέπει να υπάρχει και η καλή ασφάλιση των γυναικών, ώστε το μέλλον τους και οι συντάξεις τους να είναι εγγυημένες. Είναι σημαντικό να διευκολυνθούν οι γυναίκες οι γυναίκες συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και σε όλα τα σώματα λήψεως αποφάσεων. Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο και αυτό θα διευκολύνει τον μελλοντικό ρόλο των γυναικών στη γεωργία. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κατάσταση των γυναικών ε, στις αγροτικές ε, περιοχές εξαρτάται από την ΚΑΠ και από την κρίση. Ε, οι γυναίκες εκπροσωπούν το 40% όλων των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλειονότητα αυτών εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν πλήττονται ιδιαίτερα από το κλείσιμο των εκατοντάδων χιλιάδων μικρών εκμεταλλεύσεων και την καταστροφή των οικογενειακών αγροτικών ε, επιχειρήσεων ε, με την κοινή αγροτική πολιτική. Όλοι αυτοί οι τομείς ε, πλήττονται από την ανασφάλεια, τους κακούς μισθούς, την ανέχεια, την ανεργία. Όλα αυτά επίσης επιδεινώνονται από τις αντικοινωνικές πολιτικές. Δεν είναι λοιπόν μόνο σωστό να λέμε ωραία λόγια και να κάνουμε δηλώσεις πρόθεσης. Θα πρέπει να δώσουμε αξία στο ρόλο των γυναικών με τις πολιτικές μας και να ενισχύσουμε το δίκτυο των των δημόσιων υπηρεσιών σε αυτές τις αγροτικές περιοχές, ε, την υγεία, την παιδεία, τις οικογενειακές ε, ε, την οικογενειακή βοήθεια έτσι ώστε να μην υπάρχει η ασυμμετρία που υπάρχει στην εξοχή. Ο κύριος Νικολέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι το θέμα αυτό που έχει να κάνει με τις συνθήκες διαβίωσης ε, στις ε, αγροτικές περιοχές. Ε, πρέπει να μιλά και για τον ρόλο που παίζουν οι γυναίκες στην εξυγχρονισμό των χωριών. Επίσης θα πρέπει να ε, δοθούν τα κονδύλια της ΚΑΠ για να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ αστικών και γεωργικών περιοχών. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν εξυγχρονίζοντας ε, τις ε, υποδομές βάσης και να δώσουν υποχρεωτικά κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση. Ο αγροτικός πληθυσμός είναι σημαντικός και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν προγράμματα που θα υποστηρίζουν τους νέους εργαζόμενους στις γεωργικές επιχειρήσεις και τη δημιουργία ναι θέση εργασία για τους νέους. Η τελευταία τοποθέτηση, κυρία Νταντσίλα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Γέγκλερ για την προσέγγιση της. Νομίζω ότι η αναγνώριση του ρόλου των γυναικών στη γεωργία είναι ζωτική στην πρωτογενή παραγωγή αλλά και στην διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές και στις εκμεταλλεύσεις. Η η απομόνωση πλήττει τις γυναίκες. Χρειάζονται μέτρα αποτελεσματικά για να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες στις γυναίκες στην γεωργία ως βασικό στόχος της ΚΑΠ. Θα πρέπει να διευκολυνθούν οι συνθήκες ζωής των γυναικών που ζουν σε αγροτικές περιοχές εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην ε, συνεχιζόμενη εκπαίδευση και σε υπηρεσίες οικογενειακές. Η σημασία των ίσων ευκαιριών στις αγροτικές περιοχές προϋποθέτει καλύτερη ε, συμμετοχή των γυναικών και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες, ε, τονίζοντας τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της γεωργίας. Η κυρία Ρέντινγκ έχει το λόγο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, διότι είναι σημαντικό το θέμα το οποίο συζητήσανε και θέσανε επιτάπητος. Η Επιτροπή έχει πλήρη συνείδηση του ουσιώδους ρόλου των γυναικών στην Γεωργία και στην ε, Ήπεθρο ε, και έχουμε πολλά να κάνουμε ε, για την ανάπτυξη της αγροτικής ε, δραστηριότητας. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικούς τομείς για τις γυναίκες. Θα πρέπει να υπάρξουν μικροεπιχειρήσεις, να προσθέσουμε αξία στα γεωργικά προϊόντα και να ε, ψάξουμε για διεξόδους για την πώληση των προϊόντων τους. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης προβλέπει την βοήθεια στους άνδρες και στις γυναίκες να μπορέσουν να ε, ε, επιφέρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτική του ζωή και στις επαγγελματική δραστηριότητες. Βρεφονιπιακοί σταθμοί για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους πρέπει να υπηστηριχθούν. Επίσης, οι μεταφορές, οι μικρές υποδομές είναι επιλέξιμες για βοήθεια Έχουμε διαφορετική κατάσταση στα κράτη-μέλη, κυρίως όσον αφορά στις δυνατότητες ε, και στις απαιτήσει για τις γυναίκες. Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες πρέπει να αναλύσουν την κατάσταση και να βρούνε μέτρα κατάλληλα που συνδέονται με τις τοπικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Τα κράτη-μέλη μπορούν να δώσουν προτίμηση στις γυναίκες σε σχέση με ορισμένα μέτρα. Τα κράτη-μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς οικονομικούς για κονδύλια ούτως ώστε οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις. Επίσης οι γυναίκες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα Leader όπου μπορούν να αναδείξουν τις δυνατότητές τους για να ενεργοποιήσουν, να κινητοποιήσουν τις δυνατότητες μιας περιοχής. Η Κομισιόν συμφωνεί ότι θα ήταν πιο χρήσιμο να είχαμε περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση των γυναικών. Ωστόσο, υπό το φως της ανάγκης απλούστευσης θα ήταν δύσκολο να πείσουμε τις γυναίκες να αναλάβουν το βάρος, να αναφέρουν στοιχεία αλλά όπου είναι δυνατόν θα πρέπει να παρουσιάζονται στατιστικές και να αναλύονται αναφύλλω. Η Επιτροπή ε, θα περιλάβει στην, ε, στην έκθεσή της ε, τα στοιχεία που υπάρχουν στις κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη. Ένα σημαντικό στοιχείο σχετικά με το θέμα αυτό είναι η ανταλλαγή εμπειριών σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας πάνω στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα άλλα δίκτυα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανταλλαγή πρακτικών και θα ήταν επιθυμητό αν περισσότερες οργανώσεις γυναικών χρησιμοποιούσαν αυτά τα υφιστάμενα δίκτυα για να διασυνδεθούν οι γυναίκες στις διάφορες αγροτικές περιοχές. Ευχαριστώ Επίτροπε. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Έχει σειρά η έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου για